Ανώ, έχει το λόγο. Καταρχήν, κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε. Képviselő asszony, képviselő asszony fejezze be a kiabálást, és tisztelje meg a... Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε να φωνάζετε. Λίγο σεβασμό προς το κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ πολύ κυρία μου. Señora Presidenta. Πρόεδρε. Señora Presidenta. Usted debe proteger a los diputados. Πρέπει να προστατεύετε τους βουλευτές που έχουν το λόγο. Ε, η, μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα προσπάθησε να μπλοκάρει μια συζήτηση για τον Μπουρούντι χωρί να εξηγήσει για ποιο λόγο. Γιατί ήθελαν να διακόψουν τη συζήτηση για τον Μπουρούντι όταν εκεί στον Μπουρούντι πεθαίνουν υπέρ τη δημοκρατία. Αυτό είναι ντροπή για το κοινοβούλιο μα. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλενσιάνο. Νομίζω ότι ο καλύτερος ε, τρόπος ε, για να απαντήσουμε είναι να συνεχίσουμε μια ανιφάλια συζήτηση. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά κυρία Βαλενσιάνο. Θέλουμε να γίνουν δημοκρατικές εκλογές στον Μπουρούντι. Αλλά οι συνθήκες ε, δεν το έχουν επιτρέψει. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι εκλογέ του Μπουρούντι είναι πολύ σημαντικέ για αυτή τη χώρα, αλλά είναι σημαντικέ και για όλη την περιοχή. Θέλω να συγχαρώ τις, ε, για την εργασία της, ε, την αντιπροσωπεία μας στον Μπουρούντι, την άπατη εκπρόσωπο, τους ε, παρατηρητές μας, τον πρεσβευτή μας και τον συνάδελφο David Μάρτιν που κατόρθωσαν να αξιολογήσουν την πραγματική κατάσταση στη χώρα μια ε, κατάσταση ε, εκφοβισμού της αντιπολίτευσης, ε, απόλυτου μπλοκαρίσματος των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, μια κατάσταση μέσα στην οποία έχουν πεθάνει τουλάχιστον 40 άτομα και 100.000 άτομα έχουν διαφύγει σε γειτονικέ χώρες ως πρόσφυγες εξαιτία του φόβου. Υπεύθυνο για όλα αυτά δεν είναι κανείς άλλος από τον πρόεδρο τον πρόεδρο, ο οποίος ε, παραβίασε σαφώς τη συμφωνία της Αρούτζα, ο πρόεδρος ε, ο οποίος θεωρεί ότι η δική του προσωπική πολιτική καριέρα είναι πιο σημαντική από την ζωή και την ελευθερία των πολιτών του. Ε, το Σύνταγμα έχει καταπατηθεί, καθώς επίσης και η συμφωνία της Αρούζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στεναρή. Αν συμφωνούμε ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να ξαναβάλει ε, ε, ε, υποψηφιότητα, δεν πρέπει να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Όμως δεν καταφέραμε να συγκρατήσουμε ούτε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η Αφρικανική Ένωση την κλιμάκωση. γιατί οι κάτοικοι του Μπουρούντι χάνουν τη ζωή τους παρόλο ότι το θέμα αυτό προκαλεί το γέλιο στους συναδέλφους του EFDD, Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την οικονομική μας βοήθεια για να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών όλους αυτούς που αγωνίζονται για να γίνουν σεβαστοί, σεβαστές οι συμφωνίε τη Αρούτζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει αυτή την κοινωνία των πολιτών. Επίση, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα περιοριστικά μέτρα, να διακόψουμε τη χορήγηση θεωρήσεων, να μπλοκάρουμε ε, τους ε, λογαριασμούς της ΕΛΗ του Μπουρούντι που μπλοκάρει τις δημοκρατικέ διαδικασίε. Θα πρέπει όμω να εκφράσω και τη λύπη μου διότι ε, αν είχαν δει οι κάτι του Μπουρούντι τη σημερινή συνεδρία θα ντρεπόμασταν για την εικόνα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνθρωποι οι οποίοι παίζουν με τον κανονισμό προκειμένου να μπλοκάρουν αυτή τη συζήτηση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία. Άνθρωποι οι οποίοι φωνασκούν και περιγελούν τη συζήτηση. Αυτή είναι η εικόνα που έδωσε το κοινοβούλιο μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την υπομονή σας και ελπίζω ότι σήμερα στον Μπουρούντι γνωρίζουν, έμαθαν πως ε, παρόλο ότι κάποιοι θέλουν να διασπάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πολλοί αυτοί που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αυτών την αλληλεγγύη με τις χώρες που υποφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ταλίσκα για ένα λεπτό. Το καλύτερο παράδειγμα πολιτικής κουλτούρας ε, ε, είναι όταν ε, ζήτησα τη συνέχιση της, της ε, ε, θα ήταν να μην με αποκαλούν φασίστα και να ζητήσουν τουλάχιστον συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να σα πω το εξή για τον Μπρούντι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες. Αυτό που λείπει και παρακαλώ πολύ ενημερώστε την κυρία Μογκερίνη γι' αυτό είναι μέτρα στο πλαίσιο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ε, μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν να ασκήσουμε πίεση στο καθεστώς, στον πρόεδρο έτσι ώστε να μην χειροτερεύσει η κατάσταση. Αυτό, ε, σε αυτό δεν αναφερθήκατε στην ε, παρουσίασή σας. Παρακαλώ πολύ ενημερώστε την κυρία Μογκερίνη έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική πολιτική έτσι ώστε να ασκήσουμε πίεση στο καθεστώς. Ευχαριστώ. Ehm, Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο, για ένα λεπτό. Gracias, Presidenta. La situación de Burundi es muy grave η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και όπως πολύ συχνά συμβαίνει με την Αφρική ε, την αγνοούν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Πριν από δύο μήνες οι γειτονικέ ε, χώρες ε, υποδέχτηκαν πάνω από 100.000 πρόσφυγες που φεύγουν από την αστάθεια και την πολιτική αστάθεια και τη βία. Είναι μάθημα αλληλεγγύης για την Ευρώπη. Αυτό το οχυρό που εμένει να αρνείται το άσυλο στους γειτονές του. Ο κόσμος αιμορραγεί πολύ συχνά πια εξαιτία των συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό το λόγο το να χρησιμοποιούμε κονδύλια και τεχνική βοήθεια για να στηρίξουμε τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες ε, οργανώσεις των πολιτών επιτόπου είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι αρκετό. Τα γεωστρατηγικά ή τα εμπορικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να επικρατούν των συμφερόντων των λαών και πολύ συχνά οι πόροι της Υπήρου αυτής ε, έχουν χρησιμοποιηθεί για να αγοραστούν ευρωπαϊκά όπλα. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση στο πρόβλημα και να διευκολύνουμε το διάλογο με την ε, βοήθεια που πρέπει να δώσουμε στην Αφρικανική Ένωση. Θα πρέπει να δράσουμε υπέρ της ειρήνης. Ε, Ευχαριστώ η κυρία Σαρτζεντίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε, εμείς θεωρούσαμε ότι η συζήτηση για τον Μπουρούντι αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Πριν από δύο εβδομάδες ήμασταν έτοιμοι να μεταβούμε στη χώρα αυτή για να συναντήσουμε τους επιτόπου παρατηρητές. Και μάλιστα ε, είχαμε αρκετή ελπίδα. Φαινόταν ότι τα πράγματα θα, κάνε, θα πάνε καλά. Όμως μέσα σε μια-δυο μέρες τα πράγματα άλλαξαν από τη στιγμή που ο Πρόεδρος ε, ζήτησε να ε, έχει τρίτη θητεία. Μεσολάβησε το πραξικόπημα και εδώ που βρισκόμαστε. Στις 29 Ιουλίου θα γίνουν εκλογές αυτή την ιδέα πια δεν μπορούμε να την έχουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να την ξεχάσουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε παρατηρητές στις εκλογές αυτές γιατί θα είναι μια ε, ημέρα εκλογικής διαδικασίας εξαιρετικά βίαιη. Δεν μπορούμε να νομοποιήσουμε αυτή τη ε, διαδικασία. Αυτό που μας περιμένει λοιπόν είναι μια τεράστια κρίση με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες με οπλισμένη πολιτοφυλακή που θα υποχρεώσει τον κόσμο να ψηφίσει προς την κατεύθυνση που επιθυμεί για να παραμείνει η καθεστική ατάξη. Τι πρέπει να κάνουμε. Επίσης άλλο ερώτημα που τίθεται είναι τι ξεχάσαμε, τι δεν έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και έτσι κατέληξαν τα πράγματα εδώ που κατέληξαν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να στείλουμε αποστολή παρατηρητών στις εκλογές. Ευχαριστώ η κυρία Μακέβαν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη συμφωνία μου με την κυρία Βαλενθιάνο. Συνάδελφοι μίλησαν για το τι συνέβη στους ε, παππούς παππούδες τους πριν από 50 και 70 χρόνια στην Ευρώπη. Όμως η καταστρατηγήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασιανιστήρια, η καταστολή είναι πράγματα που συμβαίνουν εδώ και τώρα στο Μπουρούντι και γι' αυτό ε, θα μιλήσουμε. Τι θα σκέφτεται ο λαός του Μπαρούντι όταν βλέπει ότι μια συζήτηση για την τόσο σοβαρή κατάσταση στη χώρα τους ε, χρησιμοποιείται για, με φτηνά κομματικά και πολιτικά αντικατεχνάσματα από την πτέρυγα που κάθεται ε, στην, στα αριστερά μου. Η συζήτηση για το Μπουρούντι είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, έχει να κάνει με τη χώρα αυτή, με το λαό αυτό, με τους ανθρώπους που φιλοδοξούν να ζήσουν ε, σε δημοκρατικό καθεστώς. Σε δημοκρατία την οποία έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε εδώ στην Ευρώπη σήμερα. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε γιατί έχουμε μια καλή δήλωση σαφέστατη που καλύπτει όλες τις πτυχές της κατάστασης στο Μπουρούντι. Από την τελευταία σε φορά που συζητήσαμε το θέμα τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη ε, λαμβάνω από πρώτο χέρι πληροφορίες για το τι συμβαίνει, για την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τις, ε, την ένοπλη πολιτοφυλακή της νεολαίας που συνδέεται με την κυβέρνηση που κάνει φοβισμό, που ε, διενεργεί πράξεις βίας. Έχω μάθει πολλά για την Οδύνη, για το πόσο υποφέρει ο κόσμος λόγω της αστάθειας ε, στη χώρα και πόσο ε, τρέχουν να φύγουν, να σωθούν εκτός των συνόρων. Το UKIP ε, πιστεύει ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ όμως χαίρομαι διότι υπάρχει και υπάρχει και στην Τανζανία και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ε, μας θυμίσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέγας δωρητής στο Μπουρούντι. Μια χώρα η οποία είναι στη θέση 180 από τις 187 παγκοσμίω σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Τόσο πίσω λοιπόν. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε αυτή τη χώρα και δεν νομίζω ότι οι φτωχοί θα πρέπει να πληρώνουν το τίμημα της τρέλας της εκάστοτε κυβέρνησης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Μπουρούντι την ευθύνη που του αναλογεί για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει τη Συμφωνία του Κοτονού. Το Συμβούλιο υιοθέτησε σχετικά συμπεράσματα στι 18 Μαου και δεν θα πρέπει να είναι ασαφέ αυτό. Θέλουμε να γίνουν οι εκλογέ. Και θα ήθελα τέλο να ε, συγχαρώ τον David Μάρτιν, τον επικεφαλής των παρατηρητών μας. Εργάζεται εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες μαζί με τους υπολείπους συναδέλφους. Θέλουμε δημοκρατία στο Μπουρουντί και θέλουμε να γίνουν εκλογές υπό τις σωστές συνθήκες. Τα πράγματα ε, προσπαθεί να τα φτιάξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ελπίζω ότι ο κόσμος του Μπουρουντί ή τουλάχιστον η κυβέρνηση θα παρακολουθήσει τη συζήτηση στην Ολομέλεια απόψε και θα πράξει αναλόγω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπαστερετσέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγεται ότι οι βελγικές απικιακρές δυνάμεις ε, είχαν τη συνήθεια να αναφέρονται στην επικράτεια του Μπουρούντι ως Ουρούντι Ρουάντα, δηλαδή στην, ως την άλλη Ουράντα, ο άλλη Ρουάντα. Έχουμε φτώχεια, έχουμε ατιμορρησία, έχουμε έξοδο εκατοντάδων χιλιάδων. Είναι το Μπουρούντι η άλλη Ρουάντα, τίθεται το ερώτημα. Είναι μια κρίση που οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Είναι η πρόθεση του Προέδρου να παραμείνει στην εξουσία αιωνίως και γι' αυτό παραβίασε τη συμφωνία της Αρούσα. Η Ευρώπη πρέπει κάτι να κάνει. Η γενοκτονία της Ρουάντα είχε εκτός από εθνοτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Ο Γενικός Γραμματέας του του ΟΗΕ, ο Κοφεανάν, πριν από 10 χρόνια, μα είχε υπενθυμίσει την ευθύνη που είχαμε να προλάβουμε και να αποτρέψουμε αυτή τη γενοκτονία. Και στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες από τον επόμενο Γενικό Γραμματέα, τον Μπαν Κιμούν. Δεν ήταν επαρκή οι προσπάθειε. Πρέπει ε, να μην διαπράξουμε το ίδιο λάθο. Τότε δεν ε, δράσαμε εγκαίρω και υπήρξε γενοκτονία τη Ρουάντα. Τώρα, αν διαπράξουμε το ίδιο λάθο, θα είναι έγκλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, σε αυτή την αίθουσα είμαστε αναγκασμένοι και πάλι να ασχοληθούμε με την ε, οξύτατη κρίση στον Μπουρούντι. Γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε τον Ιανουάριο. Ο ένας ε, διευθυντής του ραδιοφώνου συνελήφθη και δολοφονήθηκε ε, κατόπιν είχαμε την αντικατάσταση του Προέδρου και την αναβολή των εκλογών. Αυτό οδήγησε σε σφοδρή σύγκρουση. Τα θύματα λοιπόν ήταν πάρα πολλά. Πάνω από 100.000 ήταν οι άνθρωποι που έφυγαν από τον Μπουρούντι. Όπως έχουν καταγγείλει πάρα πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ανακοινώθηκε η απόφαση του πρόεδρου Σενελίτσα να γίνουν οι εκλογές για να νεώσει την τρίτη του προεδρία. Σε αντίθεση με αυτό που προβλέπει το σύνταγμα του, ε, της χώρας. Όλοι λοιπόν πρέπει να υψώσουν αποφασιστικά τη φωνή τους και η Ευρώπη. Και είναι απαραίτητο να καλέσουμε την κυβέρνηση να επαναφέρει την κανονική, την ομαλή ε, διεξαγωγή των εκλογών με βάση αυτά που προβλέπονται στο Σύνταγμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριος Μαριάς. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Ξανά για τον Μπουρούντι. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση στον Μπουρούντι θα οδηγούσε σε συγκρούσεις η απόφαση του απερχόμενου προέδρου νκουρουτζίτζα να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία παρά τις περί του αντιθέτου αποφάσεις της συμφωνίας της αρούσα ξεχύλισε το ποτήρι. καταδικάζουμε την απόπειρα πραξικοπήματος και τις συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο μπουρούντι. ένας νέος εμφύλιος πόλεμος είναι πρώτων πυλών. πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες κατέφυγαν στις γειτονικές χώρες για να διασωθούν ο περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης πολιτικής δράσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. ήδη οι νέες εκλογές θα διεξαχθούν πλέον χωρίς τις επιβεβλημένες δημοκρατικές εγγυήσεις. η βία και οι επιθέσεις κατά των αντιφρονούντων είναι στην ημερήσια διάταξη. πρέπει λοιπόν να αναβληθούν οι εκλογές βίας και νοθείας στο μπουρούντι. για τον λόγο αυτό η διεθνής κοινότητα και η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ταυτόχρονα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να διακόψει την αναπτυσσόμενη βοήθεια στο μπουρούντι και να διαθέσει τα ποσά αυτά για τη στήριξη των προσφύγων του μπουρούντι. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσίτς. Κύριε Πρόεδρε. Το πραγματικό ερώτημα είναι μόνο ένα. Κατά πόσον τώρα βλέπουμε την αρχή του νέου εμφυλίου πολέμου κατά πόσον βλέπουμε τη δυνατότητα να επανέλθει το χάος, αλλά το χάος υπάρχει ήδη στον Μπουρούντι και υπάρχει ο κίνδυνος να μετακυλιστεί και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το ένα ερώτημα και υπάρχει και άλλο ένα ερώτημα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, τα εργαλεία με τα οποία θα μπορούσαμε να παρεμποδίσουμε επανάληψη του εμφυλίου πολέμου στον Μπουρούντι, πώς μπορούμε να αποφύγουμε, όπως σας είπα, η σύγκρουση αυτή να επεκταθεί και σε άλλες χώρες, οι οποίες επίκυνται γίνονται εκλογές. Βεβαίως και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο κύριος Μπουρουντζίζα να μην επανεκλεγεί για τρίτη φορά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουμε εκτός βέβαια αν πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες για μία τρίτη φορά, μάλλον ενός ακόμα εμφυλίου πολέμου. Στην ε, Αφρική ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακόμα ένας ε, πρόεδρος που βλέπει το τέλος της εξουσίας του προσπαθεί να αλλάξει το σύνταγμα όπως συνήθως για να παραμείνει ο αρχηγός του κράτους. Αποτέλεσμα η ξέγερση του στρατού, μερικές φορές και του λαού, πραξικόπημα ή εμφύλιος πόρεμος. Αυτή ε, είναι και η κατάσταση στον Μπουρούντι. Ε, όμως οι δημοσιογράφοι των ανεξάρτητων εφημερίδων αξίζουν την, το θαυμασμό μας. Ε, ε, ζητούν να, και, ε, και δηλώνουν ότι θα επιμείνουν παρόλη την καταστροφή ε, του press τους. Αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπεται ούτε από γεωπολιτικής πλευράς ούτε από ανθρωπιστικής πλευράς. Οι εσωτερικές ταραχές θα πλήξουν τον πληθυσμό που ήδη πεινάει. Επίτροπε, θα πρέπει να πείτε στην κυρία Μογκερίνη ότι ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, να δράσει προκειμένου να δώσει τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Ευχαριστώ. Κυρία Ρένα. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους, θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στον λαό του Μπουρούντι. Η απόφαση που ελήφθη από την Αφρικανική Ένωση να αναβληθούν οι εκλογές κατά 1,5 μήνα δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Όχι γιατί οι όροι για τη διοργάνωση των εκλογών ε, δεν πληρούνται. Ε, τα, μέ, τα μέσα μας εξενωμένως δεν υπάρχουν, ε, εκλογική δεν υπάρχει, πολυφωνία δεν υπάρχει. Θα πρέπει να εργαστούμε ε, για αυτό το θέμα και θα πρέπει να ασκήσουμε διπλωματική επιρροή αλλά και να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία. Η βοήθειά μας θα πρέπει να πάει στην κοινωνία των πολιτών και ενδεχομένως να επιβάλλουμε και ατομικές κυρώσεις, προσωπικές κυρώσεις έτσι ώστε για παράδειγμα να μην εκδίδονται θεωρήσεις για ορισμένα άνθρωπα ή να παγώσουμε ε, την, ε, τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ε, ε, ρίζα των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μποκντάνου. Α. Ε, δεν ήσασταν πριν στην αίθουσα, σας δίνω το λόγο τώρα. Κύριε Μποκτάνο, έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομο, αντίθεση με του άλλου. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι, του οποίου να του νοιάζει και πολύ το Μπουρούντι. Εγώ πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι καλούν την Ευρώπη να κάνουν τα πράγματα εκείνα τα οποία εξυπηρετούν του ίδιου Ευρωπαίου. Όταν μιλάμε για του Μπουρούντι, εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά στη τελική ανάλυση, γιατί δεν αρχίσουμε να μιλάμε για όλε αυτέ τι τηλεφωνίε ε, που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, αυτοκτονίε γιατί δεν έχουμε καλή οικονομία, γιατί έχουμε κακέ κυβερνήσει, γιατί έχουμε τόσου πολλού τους ε, μετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Γιατί δεν αρχίζουμε να μιλάμε για αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, για αυτούς που δεν μπορούμε να σώσουμε στη Μεσόγειο. Τι χρειάζεται να μιλάμε για τον Μπουρούντι. Ε, ε, μιλήσαμε για την Βερμανία. Ε, καλύτερα να μιλήσουμε για τους λαθρομετανάστες στην Ευρώπη. Μα δεν τρέπεστε να μιλάτε για αυτά που απλώς τα θέλουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μιλάμε όμως για τις επιχειρήσεις. Τι μας νοιάζει το Μπουρούντι. Εμείς εδώ είμαστε στο Μπουρούντι, μιλάμε για το Μπουρούντι, μα μιλήμαστε στην Ευρώπη. Ντρέπεστε ή δεν ντρέπεστε που μιλάτε για το Μπουρούντι. Συνάλφη, εδώ τελειώνει η διαδικασία του Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ναύρασιτς, εκ μέρους Επιτροπής. Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, ναι, χρειάζεται να στηρίξουμε το λαό του Μπουρούντι, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι τόσο καταστροφική, τόσο περίπλοκη Καταλαβαίνω και κατανοώ πολύ καλά τις ανησυχίες σας. Ε, είμαι δεκτικός εναντί των προτάσεών σας. Θα τις ε, ε, μεταφέρω στην είπατε την αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη. Όμως επειδή η κατάσταση είναι τόσο ρευστή, τόσο αβέβαιη σε ό,τι αφορά την έκβασή της, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλα τα σενάρια και όλες τις δυνατότητες ανοιχτές. Οι διαβουλεύσει ε, του άρθρου 96 Συμφωνία Κοτονού μπορούν πράγματι να είναι μία ε, δυνατότητα και άλλη δυνατότητα να ληφθούν ε, μέτρα, κυρώσει ή να δοθεί χρηματική ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση. όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένω μέτρα κοινή εξωτερική πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ε, όπως αυτά προβλέπονται και είναι διαθέσιμα ε, όπως ε, προτάθηκε από τον κύριο Ταλίτσκα. Θα πρέπει όμως να δώσουμε προτεραιότητα στην αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης και στη λειτουργία του πολιτικού διαλόγου. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τις ε, περιφερειακές ε, προσπάθειες και τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης να δημιουργήσει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για να επέλθει συμφιλίωση. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση στενά και το κάνουμε και θα το κάνουμε και θα το κάνετε και εσείς είμαι σίγουρος. Θα διατηρήσουμε την επαφή μεταξύ μας και θα επαναλάβουμε αυτό το διάλογο στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Θα ήθελα να ενημερώσω τα αξιότιμα μέλη ότι με τα λόγια του